Προέδρων έχει μοιραστεί. Δεν έχω λάβει αιτήματα για τροποποιήσει στην τελική εκδοχή τη ημερήσια διάταξη, οπότε θεωρείται αυτή εγκεκριμένη. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τώρα την εξέταση τη έκθεση τη κυρία Σακοράφα. Συμμετοχή τη Ένωση στην εταιρική σχέση στου τομεί τη έρευνα και τη κοινοτομία στην περιοχή τη Μεσογείου. Δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Σακοράφα. Panie Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σας παρακαλώ να αποχωρήσετε από την αίθουσα της Ολομέλειας ως το δυνατόν συντομότερα και θα ζητήσω την κυρία Σακοράφα να ξεκινήσει. Κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση εισηγούμε μετά από έξι μήνε εντατική αλλά ταυτόχρονα δημιουργικής συλλογικής δουλειάς της διαπραγματευτικής ομάδας της ήτρε σε συνεργασία με τη μαλτέζικη προεδρία και την ευρωπαϊκή επιτροπή την υιοθέτηση της ευρωμεσογειακής εταιρικής πρωτοβουλίας.